κυρία Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με την εντολή για τον τριγωνικό διάλογο, ο προπολογισμό του 2012, η διαδικασία καλύτερα του προπολογισμού 2012 μπαίνει στην πιο συγκεκριμένη μορφή τη. Είναι η φάση στην οποία οι αρχές του προϋπολογισμού μπαίνουν πραγματικά σε συζήτηση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμα και σημαντικά συμπεράσματα. Ελπίζω και εγώ λοιπόν ότι αυτός ο τριμερής διάλογος θα είναι μια ευκαιρία την οποία θα χρησιμοποιήσουμε και δεν θα τη χάσουμε. <clears throat> Έχουμε ξεκινήσει την άσκηση του προπολογισμού υπό την αιγίδα ενός ρεαλισμού. Τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή προχωρούν σε πολιτικές σημαντικές για παγιοποίηση και εδραίωση των προϋπολογισμών τους. Οι, οι προϋπολογιστικές αυτές πολιτικές θα πρέπει όμως να λάβουν υπόψη και την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την κρίση και να αναθερμάνουμε την οικονομία μέσω επενδύσεων. Γι' αυτό το λόγο ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει τη δική του δυνατότητα να δώσει προστιθέμενη αξία και είναι μοναδικό από αυτή την άποψη στι δαπάνε, στι επενδύσει, στου πόρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να παίξει ένα ρόλο μόχλο βραχίωνα. Είναι σημαντικό λοιπόν το σημείο αυτό και αποφασιστικό να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ως αφετηρία από τη στρατηγία του 2020. Η στρατηγία του 2020 υπεστηρίχθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη και πριν την συζήτηση επί του προπολογισμού. Γιατί ο προπολογισμό του 2012 μπορεί και θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα συγκεκριμένη δράση προ την κατεύθυνση τη στρατηγική του 2020, που είναι το μέσο το οποίο έχει επιλέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να ξαναδώσει ορμή και όθηση στις προσπάθειές μας. Το να δώσουμε μια σωστή λοιπόν χρηματοδότηση χρηματική και δημοσιονομική πτυχή στη στρατηγική του, της Ευρώπης του 2020 είναι απαραίτητο για την αξιοπιστία μας. Δεν μπορούμε να έχουμε μια τόσο φιλόδοξη στρατηγική χωρίς συγχρόνως να συνοδέψουμε αυτήν την στρατηγική με την ε, υποστήριξη που χρειάζεται για να ξεκινήσει και πάλι η ευρωπαϊκή οικονομία. Επομένως χρειάζεται συνεκτικότητα, <clears throat> αξιοπιστία για τη στρατηγική του 2020 και αυτά είναι τα θεμελιώδη στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να εξασφαλίσουμε ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε αυτή την σταθερότητα που χρειάζεται και το ενιαίο μας νόμισμα. Και έχουμε επίσης τις αναδυόμενες πολιτικές, τις ε, πολιτικές εξελίξεις στον τομέα της, χώρο της Μεσογείου, η ανάγκη να κρατήσουμε μια εξωτερική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αυτή τη στιγμή μπορεί να παίξει ένα πραγματικό ηγετικό ρόλο. Ας μην ξεχάσουμε ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι και ένα εργαλείο το οποίο έχει και χαρακτήρα προβλέψεων για τα επερχόμενα έτη. Πρέπει να λειτουργήσει λοιπόν και για το, για το τώρα και για το επόμενο χρονικό διάστημα. Επομένως, θα πρέπει να λάβει υπόψη και τα στοιχεία της εκτέλεσης του προπολογισμού του τρέχοντος για το 2011. Χρειαζόμαστε λοιπόν συνεκτικότητα, αξιοπιστία, σωστές λήψεις αποφάσεων για τον προπολογισμό, γιατί ο προπολογισμό είναι ένα θεμελιώδες εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε την κρίση και να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε τις πολιτικές λιτότητες των κρατών μελών. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα έχουμε στο νου μας και γι' αυτό έχουμε να διαδραματίσουμε ένα σημαντικό ρόλο μέσω αυτού του προπολογισμού για να εξασφαλίσουμε την σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή πρέπει να είναι η γραμμή μα κατά τη διάρκεια του τριγωνικού διάλογου. Ο τριγωνικό διάλογο θα πρέπει να είναι μια ευκαιρία για να έχουμε μια συγκεκριμένη και χρήσιμη αντιμετώπιση όλων αυτών των θεμάτων που απαρτίζουν την κοινή μας αντιμετώπιση, το κοινό μας όραμα για την Ευρώπη του 2020. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να καταλήξουμε σε κοινέ επιλογές σε αυτό το έγγραφο της εντολής για τον τριμερή διάλογο που μας δίνει την ευκαιρία να εργαστούμε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή που είναι ιδιαίτερο σημαντική και κέρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπαλτσάνη. Ο Επίτροπος κύριος Λεβεντόφσκι συνεχίζει. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Συγήτρια, Έχω έρθει για να ακούσω τις απόψει σα για το σχέδιο του προπολογισμού και την εντολή για το τριμερή διάλογο. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μα σημαντική δουλειά. Και θα έχουμε την ευκαιρία σύντομα στον επερχόμενο τριμερή διάλογο να συζητήσουμε θέματα ενδιαφέροντο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμω είναι σαφέ, και το εξήγησε και η συγκήτρια ίδια, ότι υπό τι ε, υφιστάμενε και ασυνήθει συνθήκε η σύνταξη του προπολογισμού του 2013 δεν μπορεί να είναι κάτι το συνηθισμένο, δεν μπορεί δηλαδή να ακολουθήσει τα ιωθώτα έτσι, θα πρέπει και να ε, είναι σωσκελισμένος ο προϋπολογισμός αλλά και να δίνει ενίσχυση και υποστήριξη στην ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Είναι σαφέ νομίζω από το σχέδιο, γιατί ακόμη και την ε, στιγμή της κρίσης χρειάζονται επενδύσεις για να βοηθήσουμε την πολύ ευάλωτη οικονομία της Ευρώπης να ανακάμψει. Αυτή είναι η απάντηση λοιπόν που μπορούμε να δώσουμε καταρχάς στο σχέδιο αυτού του προπολογισμού. Επίσης έχουμε σε φως αναβαθμίσει τις ε, προτεραιότητες για την ε, στρατηγική για την Ευρώπη 2020 62,6 δισεκατομμύρια, δηλαδή 43,5% του σύνολου του σχεδίου προϋπολογισμού. Αναβαθμίζουμε επίσης τις ε, δαπάνες που σχετίζονται με τη συνθήκη της Λισαβόνας το 4, κατά 4% και έχουμε μια πολύ αυστηρή προσέγγιση στα θέματα της ε, γραφειοκρατίας, της διοίκησης, δηλαδή με μηδενική αύξηση στον τομέα της Επιτροπής και με πολύ αυστηρή εξέταση των επιδόσεων και της εργατικότητας του προσωπικού. Είναι πολλές φορές ε, χαμηλότερη χρηματοδότηση από τις υφιστάμενες ε, προοπτικές του 2000, από το υφιστάμενο προϋπολογισμό του 2012. Και λησμονούμε ότι ο προϋπολογισμός του 2012 ήταν 9 δισεκατομμύρια χαμηλό, κατά 9 δισεκατομμύρια χαμηλότερος από αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί στο σχέδιο. Όταν βλέπουμε ένα σχέδιο προπολογισμού, έχουμε την υποχρέωση βέβαια, ε, εξετάζοντά τον, να δίνουμε απάντηση στα παγκόσμια προβλήματα. Εν προκειμένου την τι εξελίξει στη Μεσόγειο. Και γι' αυτό έχουμε την πρώτη ορθωτική επιστολή για τον προπολογισμό τη προηγούμενη εβδομάδα, που στόχο έχει να αναβαθμίσει τη δημοσιονομική ανταπόκριση στα θέματα τη γειτονία και ιδιαίτερα την όχθη τη Μεσογείου, αυξάνοντα κατά 1 δι 300 εκατομμύρια το, ποσοστό, το ποσό που θα διατεθεί και έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα για, την άμεσο, για το άμεσο διάστημα που ακολουθεί να ε, διοχετεύσουμε 500 εκατομμύρια ε, στις ε, χώρες της Όφης Μεσογείου και την ευρύτερη γειτονία μέσω των μέσων ευελιξίας με 153 εκατομμύρια ευρώ ιδιαίτερος. Το αποτέλεσμα είναι σαφές, ε, παρουσιάστηκε άλλωστε, θα έχουμε αύξηση στις πληρωμές κατά 4 περίπου της 100, όχι όμως ε, μεμονωμένη. Στόχο έχει ιδιαίτερα να καλύψει τις υφιστάμενες ε, νομικές υποχρεώσεις και για να επαναλάβω άλλη μία φορά, 9 δις ή μάλλον 8,8 για να είμαστε πιο ακριβείς δισεκατομμύρια, χαμηλότερα από αυτά που είχαν προβλεφθεί στο ανώτατο επίπεδο, προφανώς σημαίνει ότι μας λείπουν πόροι από τον, το φετινό, από τον προπολογισμό του 2012. Τώρα έχουμε κάποιες υποχρεώσεις οι οποίες είναι λεξιπρόθεσμες και πρέπει να καταβάλουμε τα σχετικά ποσά. Ακόμη και έτσι η αναβάθμιση είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή που προβλέπεται στους αντίστοιχους προπολογισμού για τα κράτη-μέλη ε, του 2012. Δεν βλέπω ότι θα είναι ε, πολύ εύκολη συζήτηση με το Συμβούλιο. Άλλωστε έχουμε και ε, το παρελθόν που δείχνει κάποια στάση, δηλαδή τον προπολογισμό του 2012 και έτσι περιμένει υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να έχουμε και έναν καλά ισοσχελισμένο προπολογισμό αλλά και επαρκή επενδύσει και ανάπτυξη για ε, τον ε, προπολογισμό του 2013 με την ελπίδα ότι θα είναι η διαδικασία λιγότερο ταραχώδης και έντονη από αυτήν του προπολογισμού του 2012. Ευχαριστούμε. Κύριε Επίτροπε, για 1,5 λεπτό τώρα εκ μέρου τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, η κυρία Μουνή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο προπολογισμό του 2012 λένε ότι πρέπει να περιοριστεί στα αναγκαία προκειμένου να καλύψει τι νομικέ υποχρεώσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμω τι σημαίνει. Σημαίνει να παγώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμεί δεν συμφωνούμε. Στην Ευρώπη εμεί ε, θέλουμε τι πολιτικέ τη, συμφωνούμε με αυτέ και θέλουμε να εκτελεστούν. Δεν πρόκειται για δαπάνε, πρόκειται για πρόσθετη αξία. Όπω λέει και η συγγήτρια, ε, συμφωνούμε και εμείς για το ότι ο προπολογισμό πρέπει να προσανατολίζεται στη στρατηγική 2020 υπέρ τη ανταγωνιστικότητας και τη απασχόλησης. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να χάνουμε από μπροστά μας ε, την υποχρηματοδότηση διάφορων δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο Θέλουμε μαζί να φροντίσουμε η Ευρώπη να αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα με το 2,9% ναι που δεν έκανε ο πληθωρισμός. Η πρόταση που γίνεται σήμερα δείχνει τη βούλησή μας να προωθήσουμε την ειρήνη, την ανάπτυξη και τη διεθνή σταθερότητα, όπως επίσης και τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο. Θα επικεντρωθώ εγώ στα σημεία τα οποία απασχολούν περισσότερο την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Πρώτα απ' όλα, η επαναδιατύπωση της πολιτικής γυτνίασης με τη μεσογειακή της διάσταση πρέπει να χρηματοδοτείται επαρκώς από τον προπολογισμό. Και για να ξεκινήσουμε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την Παλαιστίνη και την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και την δεν χρηματοδοτείται επαρκώς, αντίθετα πλήττεται με μια μείωση των 100 ε, εκατομμύριων ευρώ. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο και η δουλειά της UNRWA είναι πάρα πολύ σημαντική για να μειώσουμε την χρηματοδότησή μας χρόνο το χρόνο. Μειώνει η Κομισιόν τα ποσά κάθε χρόνο και μετά βέβαια γίνεται η γνωστή διαπραγματεύση στον προπολογισμό. Έπειτα, η Μεσόγειο είναι πολύ σημαντική, κύριε Επίτροπε, αλλά όχι σε βάρο άλλων διαστάσεων τη εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, Λατινική Αμερική, που και αυτή δεν χρηματοδοτείται επαρκώ ιστορικά. Κάτι που σημαίνει ότι μπλοκάρουμε τελικά τα ποσά από χώρε οι θα μπορούσαν να αποφελεθούν. Και ολοκληρώνω, Πρόεδρε. Δεν γίνεται αυτό επειδή βρίσκουμε κάποια λύση στη νομική βάση. Όχι, η διεύρυνση και το ο μηχανισμό σταθερότητα πρέπει να προχωρήσουν. Και κάτι για τα πολυμέρη, όπω η συνεισφορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι γυναίκε. Δώστε μου μισό δευτερόλεπτο, Πρόεδρε. Πρόκειται επίση για το να χρησιμοποιούμε βέλκτα τον προπολογισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού για ένα λεπτό, ο κύριος Χατζημαρκάκης. Κύριε Πρόεδρε, από την οπτική γωνία της Επιτροπής Ελέγχου του προπολογισμού, πολλές φορές υπάρχει η εντύπωση ότι υπάρχουν πραγματικά προβλήματα στην εκτέλεση του προπολογισμού, ατασταλίε κτλ. πάντα, αλλά πρόκειται κυρίω για τα κράτη-μέλη τα οποία είναι υπεύθυνα για τα θέματα αυτά και που έρχονται με τον κύριο Κάμερον τα κράτη-μέλη και λένε τι μας, γιατί μας ζητάτε περισσότερα λεφτά, πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε καλύτερα. Ενώ αυτή είναι υπεύθυνη. Και το 2010 ποιος ήταν ο χειρότερος φταίχτης στα θέματα αυτά, η Μεγάλη Βρετανία πολλά από τα βρετανικά προγράμματα ουσιαστικά σταμάτησαν στη, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ πολύπλοκοι οι κανόνε. Γι' αυτό θέλω να ζητήσω από την Κομισιόν να μπορέσει να συζητήσει με τα κράτη μέλη για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε απλούστερα συστήματα, απλούστερα συστήματα ελέγχου και να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια ε, ανταμοιβή κατά κάποιο τρόπο για αυτούς οι οποίοι έχουν πραγματικά καινοτόμα και σημαντικά προγράμματα και το ίδιο θα πρέπει να συμβεί σε προγράμματα που είναι στον τομέα της ε, συνοχής που μπορούν να παίξουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα αυτά τα αποτελέσματα. Μπορούμε λοιπόν με τον τρόπο αυτό να ευνοήσουμε μια ανανέωση και μια καινοτομία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Χατζημαρκάκη. Από την Επιτροπή Απασχόλησης για ένα λεπτό κύριε Μπερές. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Οι προτεραιότητες που όρισε η Επιτροπή των Κοινωνικών Υποθέσεων εκείνων από μια ανησυχητική διαπίστωση ότι εξακολουθεί να μένεται η μεγάλη οικονομική κρίση. 28 εκατομμύρια άνεργοι με 5,2 νέους εκατομμύρια. Και έτσι λοιπόν η πολιτική για την απασχόληση των κρατών μελών θα έπρεπε να διαμορφωθεί κατά τρόπον ώστε όπως και το Κοινοβούλιο από το Συμβούλιο να μην θεωρεί ως δευτερεύον μέτρο και δευτερεύουσα διάσταση της ανάπτυξης στην απασχόληση θα έπρεπε να γίνει μεγάλη προτεραιότητα για την περίοδο 2011-2012. Πρόκειται για μια ε, διεκδίκηση την οποία θα πρέπει και ο προπολογισμό να εκφράσει υποστηρίζοντας τους πέντε μεγάλους στόχους της ε, στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 και ειδικότερα το ημείωση του ποσοστού εκείνων που πλήττονται από την φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό και την αύξηση του ποσοστού της απασχόλησης συμπληρωματικότητα, αναλογικότητα και συγκρισιμότητα μεταξύ του προπολογισμού και των μέτρων που εφαρμόζονται. Ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια κυρία Μπαλτσάνη, γιατί ξέρουμε ότι στον τριμερή διάλογο υποστηρίζει ιδιαίτερο τι θέσει τη Επιτροπή Απασχόληση. Ευχαριστούμε. Εκ μέρου τη Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη, για ένα λεπτό έχει το λόγο ο κύριο Σούζαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης πρέπει να σας πω ότι συζητήσαμε και εγκρίνουμε την πρόταση. Πιστεύουμε ότι προετοιμάστηκε ιδιαίτερα προσεκτικά προκειμένου να προετοιμαστούμε για τον τριμερή διάλογο και προκειμένου να προχωρήσει καλά η δημοσιονομική διαδικασία. Για την Επιτροπή μας το στοιχείο κλειδί είναι η χρηματοδότηση της πολιτική συνοχής. Θέλουμε λοιπόν να υπογραμμίσουμε ότι Κατά τη διάρκεια του 7 δημοσιονομικού κύκλου έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου τα κράτη-μέλη περιορίζουν τα ιδιαίτερα ψηλά ε, ποσά, μεγάλα ποσά, από την άλλη μεριά όμως εξοδεύουν περισσότερα. Η κατάσταση λοιπόν έχει ως εξή. Πέρυσι το διπλάσιο ποσό δαπανήθηκε από ό,τι οποιαδήποτε προηγούμενη χρονιά. Αυτό τι δείχνει. Δείχνει ότι υπάρχει επιτάχυνση, υπάρχουν βέβαια και εθνικοί λόγοι, γιατί υπάρχουν και διάφορες τάσεις σε πολλές χώρες, όχι μόνο σε μία. Ελπίζω να στηρίξετε την πολιτική αυτή. Ευχαριστούμε κύριε Σιουζέν. Εκ μέρους της Επιτροπής Γεωργίας τώρα για ένα λεπτό έχει το λόγο ο κύριος Κάπουλας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για το δεύτερο τίτλο, κοινή αγροτική πολιτική, τρία βασικά θέματα. Για τον πρώτο πυλώνα δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, δεδομένου του ότι 90% των δαπανών βρίσκονται στον τομέα αυτό και η εκτέλεση, η απορρόφηση είναι περίπου 100%. Το 2012 υπάρχει μονάχα μια τροποποίηση κατά 3% των κονδυλίων για να προσαρμοστούν στο κόστος της διεύνησης. Ούτε και ο δεύτερος πυλώνας δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα γιατί και εκεί υπάρχει μια αύξηση των ε, δαπανών ως τμήμα της ε, πορείας της ε, δημοσιονομικής περίοδου προγραμματισμού και αυτό είναι θετικό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της διεύρυνσης. Ο τρίτος τώρα πυλώνας είναι αυτός ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει ορισμένα προβλήματα. Τα προγράμματα διανομής φρούτων και λαχανικών στα σχολεία και επίσης αυτά τα οποία μειώθηκαν ιδιαίτερα μετά από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου γιατί ο στόχος ήταν να υπάρξει κινητοποίηση κονδυλίων για να μπορέσουν να διανεμηθούν και να αξιοποιηθούν πλεονάσματα μέσω του μηχανισμού αλληλεγγύης. Και η αλληλεγγύη δεν πρέπει να είναι μονάχα ένα σύνθημα πολιτικό, πρέπει να είναι κάτι το οποίο πριτανεύει στην συνείδηση της ε, Κομισιόν και του Συμβουλίου όταν κάνουν προτάσεις και πρέπει να κάνουν προτάσεις να διορθώσουν αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάπουλος για την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων για ένα λεπτό ο κύριος Λούντβιγκ Σον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Από την πλευρά της Οικονομικής Επιτροπής εγώ θα ήθελα να θίξω τρεις προτεραιότητες. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει οι νέες εποπτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τύχουν τη σωστή χρηματοδότηση θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να εργάζονται σωστά και στεναρά για το καλό των χρηματοπιστωτικών αγορών. Πρέπει να έχουμε επίσης τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε τη σωστή και επαρκή στελέχωση σε προσωπικό αυτών των υπηρεσιών. Επίσης, στα θέματα τα οικονομικά πρέπει και η ίδια η Κομισιόν να ενισχύσει τις δομές της και από τη στιγμή θα πρέπει να υπάρξουν σωστές ρήτρε ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν με αποτελεσματικό τρόπο και αυτό απαιτεί και βελτίωση των στατιστικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί οι ανεπαρκείς στατιστικές είναι και αυτές αιτία για την κρίση. Ευχαριστώ για την Επιτροπή Βιομηχανίας και για ένα λεπτό ο κύριος Κόφερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Συγγετρία. Καταρχά ευχαριστώ εξ ονόματο τη Επιτροπής μα ε, θερμά την εισηγήτρια. Ήταν πολύ εντατική και πολύ θετική η στάση τη στην ε, συνεργασία και πρέπει να σημειώσω δίνει το καλό παράδειγμα με τη συμπεριφορά αυτή. Κύριε Επίτροπε, είπατε ότι δεν πρέπει να ακολουθήσουμε την πεπατημένη. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Και αν σας έλεγα ότι οι προτεραιότητες οι ενεργειακές Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Στρατηγικής 2020 ε, έχουν προσδιοριστεί όπως έχουν προσδιοριστεί και τις συγκρίνουμε αυτές με τις προτάσεις της Επιτροπής, μάλλον ακολουθεί τα ιωθώτα η Επιτροπή, διότι δεν δίνει επαρκή χρηματοδότηση και μάλιστα προβλέπει και περικοπές σε σημαντικό τομέα της ε, ενέργειας. Όπως λένε οι Αμερικανοί, we must put our money where our mouth is. Αυτά που λέμε δηλαδή και να τα χρηματοδοτούμε. Ε, πράγμα το οποίο δεν κάνετε εσείς. Επίσης η Επιτροπή Βιομηχανίας ανησυχεί διότι υπάρχει μια εκρηκτική αύξηση σε δαπάνες ε, στο ΙΤΡ και στο ΠΑΕΣ που όμως δεν αντισταθμίζεται από δαπάνες υψηλές και στην έρευνα. Αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να ολοκληρώσω θέλουμε προτεραιότητες για την πρόσβασή τους στα μέσα καινοτομία, στα μέσα της έρευνας και, στην καινοτομ... και στην... Ε, στους μηχανισμούς καινοτομίας. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους των πολιτικών ελευθεριών. Η κυρία Κέλλερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή Ελευθεριών του Πολίτη χαίρεται πολύ για την ε, αύξηση στον τομέα της δικαιοσύνης και ελευθεριών του πολίτη. Χρειάζονται νέα προγράμματα και να αξιολογηθούν καλά τα τρέχοντα. Οι αξιολογίες αυτέ πρέπει να ληφθούν ω βάση για την εκπόνηση νέων προγραμμάτων. Υπάρχει περιθώριο λοιπόν για συνέργειε, για να αποφεύγουμε επικαλύψεις και να γίνουν τα πράγματα απλούστερα, έτσι ώστε να προσφέρουμε μια προστιθέμενη αξία με ό,τι κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή μας πιστεύει ότι πρέπει να κοιτάμε καλά τι συμβαίνει γύρω μας σήμερα, τη συγκεκριμένη στιγμή και ανάλογα να φροντίσουμε για τις δαπάνες μας, για την προστασία των πολιτών αλλά και για την ένταξη των Ρώμα. Όλες οι υπηρεσίες μας, όλοι οι οργανισμοί μας πρέπει να φέρουν σε πέρας ε, τα καθήκοντα τα οποία έχουν αναλάβει. Και τέλος, και μπορεί να ενδιαφέρει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό, η Επιτροπή μας πιστεύει ότι ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού πρέπει να πηγαίνει στο αποθεματικό, μια που δεν υπάρχουν ακόμα αποτελέσματα και ένα μέρος των δαπανών για το προσωπικό επίσης θα το βάλουμε στο αποθεματικό στην περίπτωση που δεν δούμε να παρουσιάσετε το UFTT το πρόγραμμα το οποίο περιμένουμε από την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Κέλλερ. Ο κύριος Αντάργας δεν είναι εδώ από ό,τι βλέπω. Δεν είναι στην αίθουσα. Οπότε, για ένα λεπτό, εκ μέρους της Επιτροπής Δικαιωμάτων της Γυναίκας, το λόγο έχει η κυρία Ματέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ευαίσθητο το πλαίσιο το χρηματοοικονομικό και δημοσιονομικό στα κράτη-μέλη και δείχνει ότι δεν επαρκεί στι προσπάθειε των ευρωπαϊκών χωρών για να αντιμετωπίσουν την κρίση του δημόσιου χρέου. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει σε κέριου τομεί μία μείωση των επενδύσεων και μία μείωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η στρατηγική 2020 που είναι το κέντρο του προϋπολογισμού του 2020 προτείνει να υπάρχει μία οδός η οποία πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά και αντιμετωπίζει με την ε, ευθύνη της ε, Κομισιόν για να υπάρξει η αντιμετώπιση του, της στρατηγικής 2020 αλλά συγχρόνω δεν μα ικανοποιεί το γεγονό ότι μειώθηκαν τα κονδύλια σε προγράμματα όπω το Progress που έχει μεγάλη σημασία για να βοηθήσει την απασχόληση των νέων και να αντιμετωπίσει την ένδυα και να εξάρει την ισότητα των ε, φίλων. Επίση, το πρόγραμμα Δάφνη, το οποίο έχει σαν στόχο να αντιμετωπίσει τη βία κατά των γυναικών, είναι απαραίτητο να τύχει σωστή χρηματοδότηση. Γι' αυτό θέλουμε ο προπολογισμό του 2012 να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουμε πιο συγκεκριμένο τρόπο τι προκλήσει που έχει ενώπιον τη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ κύριε Ματέρα. Περνάμε στους ομιλητές εξορμός των πολιτικών ομάδων για την ομάδα του ΕΛΚ. Δύο λεπτά. Ο κύριος Λαβία. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τα τρία κύρια θεσμικά όργανα μέσα στα πλαίσια του προπολογισμού έχουν να αντιμετωπίσουν ένα δύσκολο εγχείρημα πρέπει να φτάσουν να έχουν ένα επίπεδο πόρο στον προπολογισμό που λαμβάνει υπόψη τι προκλήσει που έχει ενώπιον τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί από τα προηγούμενα χρόνια. Θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία σε σχέση με την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντα με απόλυτη επίγνωση να υπάρξει μια λιτότητα αλλά σε επίπεδο ευθύνη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να ψηφίσει αυτό το σημαντικό έγγραφο το οποίο είναι η εντολή για τον τριμερή διάλογο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο το ΕΛΚ θέλησε να ενισχύσει το έγγραφο αυτό της εισηγήτριας κυρίας Μπαλτσάν, την οποία φυσικά υποστηρίζουμε και ευχαριστούμε για τη θαυμάσια εργασία της και θέλει το ΕΛΚ θέλει να τονίσει τη σημασία του να υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι για τη χρηματοδότηση των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 που βρίσκεται στην καρδιά, στον πυρήνα του προϋπολογισμού του 2012. Είναι σαφές ότι μόνο με τη βοήθεια του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού θα μπορέσει να αντισταθμιστεί η έλλειψη πόρων στα εθνικά κράτη. Χρειάζεται να υπάρξει λοιπόν αηφόρος ανάπτυξη, υποστήριξη στην καινοτομία, στον τομέα της εργασίας, στη μεγαλύτερη απασχόληση και κυρίως για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όλες αυτές είναι οι προτεραιότητε μας. Πιστεύω ότι οι επενδύσεις στους τομείς αυτούς είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσει η Ευρώπη να βγει από την κρίση. <clears throat> Υποστηρίζουμε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτή η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσα από τον προϋπολογισμό και την δημοσιονομική σχεδίαση. Υπάρχει μια... Ε, ένα ακόμα σημείο. Θέλω να τονίσω την ανάγκη να μην γυρίζουν οι πόροι οι οποίοι δεν έχουν δαπανηθεί στα κράτη-μέλη, αλλά να παραμένουν στον προϋπολογισμό. Να υπάρχει η ρήτρα νήσιν αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το πλαίσιο το οποίο επιτρέπει στην Κομισιόν να κάνει κάτι τέτοιο. Νομίζω και ότι αυτό πρέπει να γίνει και επίσης σας λέω ότι δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα προβλήματα του προηγούμενου Δεκεμβρίου θα πρέπει ήδη από, την, από τον τριγωνικό διάλογο του Ιουλίου να έχουμε μια ισορροπία στις διαπραγματεύσεις μέσα στα κάτι μέλη χωρί να παραγνωρίσουμε τι στρατηγικές προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίε είναι απαραίτητε για την αναθέρμανση τη οικονομία τη Ευρώπη και για τα 520 εκατομμύρια πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρου των Σοσιαλιστών. Πάνω στην ώρα. Για ένα μισή λεπτό έχει το λόγο η κυρία Χέρτσοκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, έφτασα άγκαιρα. Και καλημέρα σε όλους σας. Ο προπολογισμός για το 2012 είναι ο μικρός αδερφός του πακέτου οικονομικής διακυβέρνησης. Οι στόχοι είναι λίγο πολύ το ίδιο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για οικονομική και δημοσιονομική ισορροπία, να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, χρησιμοποιώντας ε, τα κατάλληλα δημοσιονομικά μέσα. Χρειαζόμαστε αποτελέσματα, χρειαζόμαστε θέσεις απασχόλησης, χρειαζόμαστε ανάπτυξη, χρειαζόμαστε βιομηχανική πολιτική, με άλλα λόγια χρειαζόμαστε μια ισχυρή ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε αύξηση του ΑΕΠ κάτω από τις συνθήκες που βρισκόμαστε σήμερα. Έχουμε ένα σταθές ευρώ. Άρα πώς είναι δυνατόν τα κράτη-μέλη να έχουν καλύτερες επιδόσεις και να αυξήσουν το ΑΕΠ Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξυπηρετεί τους πολίτες της. Γι' αυτό και θέσαμε στόχους και πρέπει να συνεχίσουμε με την στρατηγική 2020. Αντί για ύφεση, η Ευρώπη πρέπει να έχει ηγετικό ρόλο στην καινοτομία. Χρειαζόμαστε μια νέα βιομηχανική επανάσταση. Ο προπολογισμό για το 2012 πρέπει να αποτελεί μέρος της στρατηγικής 2020. Μιλάμε για τη δεύτερη χρονιά του δεκαετούς αυτού προγράμματος. Δεν μπορούμε λοιπόν απλώς να πούμε ότι θα δώσουμε αποτελέσματα αργότερα τα 17 χρόνια. Δεν μπορούμε τώρα να γυρίσουμε και να πούμε στους πολίτες ότι θα κάνουμε περικοπές στον προπολογισμό. Ο προπολογισμός για το 2012 και το 2013 πρέπει να ικανοποιήσουν τις ανάγκες αυτές. Ευχαριστούμε για δύο λεπτά τώρα ο κύριος Χάκλουν επέρους των φιλελεύθερων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω το, την εξαίρετη ε, δουλειά για την εξαίρετη δουλειά την ε, εισηγήτρια. Η στρατηγική 2020 αποτελεί το μυαλό τη στην υπόθεση αυτή. Είναι μια στρατηγική δηλαδή που μας στρέφει προς το μέλλον, μια στρατηγική με την οποία εγγράφονται και γράφεται και το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο και πιστεύω ότι ο προπολογισμό του 2013 θα έχει καθοριστική σημασία εν προκειμένου. Έχουμε ξεκινήσει μια μακρά και δύσκολη διαδικασία ήδη από τον προπολογισμό του 2011 όπου μπορέσαμε με δυσκολία μόνο να βρεθούμε στο ίδιο με το Συμβούλιο. Και πρέπει να εκφράσουμε δυστυχώς ε, τη λύπη μας για ορισμένε από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2012. Υπάρχουν προτάσεις οι οποίες ε, είναι υπερβολικές κατά την έποψή μας. και πιστεύω ότι θα πρέπει αντί να αυξάνονται τα ποσά να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα. Είναι ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε. Και ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι κάθε χρόνο σε τομεί τομείς όπου ζητάμε ε, επιπλέον ζητούνται επιπλέον ποσά ε, ότι δεν υπάρχει επαρκής απορρόφηση και σωστή διαχείριση. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Δεν μπορεί να είναι ο προπολογισμό διωγγωμένο όπω τον ζητεί η Επιτροπή, χωρί αποτέλεσμα. Είναι σαφέ ότι δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε μηδενική ανάπτυξη, έστω. Αλλά οι προτεραιότητε πρέπει να διαφοροποιηθούν, πρέπει να οριστούν κατά καλύτερο τρόπο. Και η ομάδα μας θα μπορεί τότε να αναλάβει τι ευθύνες της, αλλά μόνο όταν είναι και υπεύθυνη η, η σύσταση του προπολογισμού. 1,5 λεπτό ο κύριος Μπόκρος. Έχει πτωχεύσει το ελληνικό κράτος. Το θέμα δεν είναι μόνο η συγγνώμη, αλλά ακόμα και συγγνώμη όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο. Πρέπει να καταλάβουμε τη φύση του προβλήματος όμως η χρόνος. Δεν είναι θέμα ρευστότητα, αλλά είναι ένα θέμα βαθιάς φαρεγγιότητας που δείχνει ότι υπάρχει έλλειψη ανταγωνιστικότητα από πλευρά τη ελληνική κυβέρνηση. Το να βάζουμε να πληρώσουν περισσότερου φόρου οι Έλληνε είναι αντιπαραγωγικό. Το να αρχίσει, για να αρχίσει να ε, βγαίνει από το χρέο η Ελλάδα πρέπει αυτό να φύγει, να συγχωρεθεί και να ξεκινήσει η ιδιωτική πρωτοβουλία. Για τις ελληνικές τράπεζες πρέπει να υπάρξει κεφαλοποίηση. Η, τα ομόλογα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την πολιτική της μέχρι τώρα έχει βρεθεί σε παγίδα. Ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα χρειάζεται η οποία να απαγορεύει την κεφαλοποίηση του δημοσίου χρέους. Χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων και τώρα πληρώνουμε τις συνέπειες και ακριβώς αυτά τα πλαίσια πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τον προϋπολογισμό για το 2012. Είναι ψευδέστηση να περιμένουμε ανάπτυξη ε, και περισσότερη συνεισφορά των χωρών μελών στον προπολογισμό αυτό. Δεν είναι δυνατόν. Οι επιστολές των πρόεδρων και των πρωθυπουργών των πέντε χωρών πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι, μην τις ξεχνάμε. Έχει αποτύχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρυσι και πρέπει και αυτό να το θυμόμαστε. Η εντολή για τον τριμερή διάλογο πρέπει να είναι πιο μετριοπαθής και πιο ρεαλιστική εφόσον επιθυμούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παραμείνει να έχει νόημα για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπόκρε. Από τους Πλασίνους, ε, Ελεύθερη Συμμαχία, για ένα λεπτό κυρία Τρίπελ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα καταρχάς να υποστηρίξω εν γέννη όσα είπε ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι, ότι δηλαδή σε περίοδους κρίσης χρειάζεται να εξισορροπηθεί η αναγκαία βεβαιολιτότητα αλλά και η αξιοποίηση και η, η αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά ταυτόχρονα και οι ε, επαρκείς σπόροι οι οποίοι δεν θα υποβαθμίσουν τις οικονομικές μας δυνατότητες. Αυτές είναι οι κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες συμμερίζομαι και που πιστεύω ότι θα πρέπει να αποτελήσουν το μέτρο για τον προϋπολογισμό μας. Πλην όμως, αυτή η πρόθεση, η σωστή αυτή προσδοκία την οποία ορίζει και περιγράφει ο Επίτροπος υλοποιείται το όντι μέσα σε αυτή την πρόταση. Εμείς ως πράσινοι θεωρούμε ότι δεν ισχύει αυτό. Όταν έχουμε επί παραδείγμα την περίπτωση του αντιδραστήρα ΙΤΕΡ ως εγχείρημα το οποίο έχει τη μεγαλύτερη αύξηση κονδυλίων με 740 εκατομμύρια ευρώ από, από τον ολόκληρο προπολογισμό, αμφισβητούμε το κατά ορθή επιλογή σε τέτοιε εποχέ, όταν άλλα ε, σχέδια, οι Φερρυπίν και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βλέπουν ε, την ε, χρηματοδότηση τους να μειώνεται. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αποτελούν από ό,τι φαίνεται προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μόνο το ίτερ. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι λάθος οι επιλογές σας προς προτεραιότητες και δεν θα τις μεριστούμε. Ευχαριστώ κυρία Τρίπελ <coughs> για την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, πράσινη σκανδιναβική αριστερά. Για ένα λεπτό κύριο Πόρτας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο. Η ομάδα μου συμφωνεί με την εντολή διαπραγματεύσεως με το Συμβούλιο που θα εγκρίνουμε σήμερα, αλλά θα ήθελα να θέσω ένα πολιτικό θέμα το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο έγγραφο αυτό <clears throat> και έχει να κάνει με την κατάσταση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και η δική μου χώρα η Πορτογαλία. Και με τις δηλώσεις του Jean-Claude Juncker. Οι δύο αυτές χώρες και κατά πάσα και άλλες χώρες στο μέλλον θα αντιμετωπίσουν ένα φαύλο κύκλο πολιτικών διάσωση. Η μία διάσωση θα σώσει την προηγούμενη διάσωση. Αυτή η κόλαση που προέρχεται από την πολιτική λιτότητα έχει σαφείς επιπτώσεις για και οδηγεί σε μείωση του επίπεδου δημοσίων επενδύσεων και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Είναι απαραίτητο λοιπόν το 2012 και το 2013 η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε θέση να έχει μια πολιτική σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των διαφορετικών ταμείων για τις συγκεκριμένες αυτές χώρες που να μην δίνει μονάχα προκαταβολές σε ό,τι αφορά τα ταμεία αυτά που θα καταβληθούν, αλλά και συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να μειωθεί η συγχρηματοδότηση από τα εθνικά κράτη για τις ε, επενδύσεις που είναι παραγωγικού χαρακτήρα και προωθούν την ε, απασχόληση. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα δύο χρόνια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πόρτας για την ε, Ευρώπη της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας. Για ένα λεπτό κύριε Αντρίεσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ενώ συζητούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διασωθεί η Ελλάδα από τη χρεοκοπία, χρεοκοπία η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλη οικονομική ύφεση και δημοσιονομική σε ολόκληρο τον κόσμο, συζητούμε μια αύξηση του προπολογισμού μας κατά, κατά 5% για το 2012. Αυτό που αποτελεί ασφαλμένο μήνυμα για τους πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Δεν ενισχύει την αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ευρωπαϊκός προπολογισμό δεν θα μας βγάλει από την κρίση, ούτε και μπορεί να μας βγάλει από την κρίση. Υπάρχουν διάφορα τμήματα του προπολογισμού που όλοι γνωρίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε Περιπλο- περικοπές. Πρέπει να σταματήσουν τα ε, σχέδια και τα προγράμματα τα οποία δεν έχουν φέρει αποτελέσματα. Πρέπει εκεί όπου δεν υπάρχει σωστή αντιμετώπιση των ε, δικαιωμάτων των πολιτών σε διάφορες περιοχές όπου υπάρχουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων να διακοπεί η χρηματοδότηση και αυτή θα πρέπει να είναι η γραμμή που θα χαρακτηρίσει τον προπολογισμό του 2012. Εάν αυτό δεν συμβεί, τότε θα καταλάβουν οι πολίτες ότι μόνο η αρχική των κρατών και κυβερνησεών τους θα μπορέσουν να τους υπερασπιστούν. Ευχαριστώ πολύ για μέρους των μη εγγεγραμμένων και για ένα λεπτό. Ο κύριο Χάρτουγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα μιλάμε για τον προπολογισμό του 2012. Η ομάδα μα είναι κατά των προτάσεων που γίνονται για αύξηση 5%. Είναι μια πρωτοβουλία που δεν μπορεί να βοηθήσει, γιατί δεν είναι δυνατόν να ζητάμε χρήματα από τους Ευρωπαίους για να πληρώνουν οργανισμούς που δεν λειτουργούν. Και για τις λεπτομέρειες, 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ απαιτούνται για το ΙΤΕΡ. Πολλά χρήματα, τα οποία πρέπει να τα πάρουμε από αλλού βέβαια. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται αναθεώρηση. Κάθε κράτος μέλος όμως έχει βέτο, αρνησικυρία για τον προπολογισμό το 2012. Πάρα πολύ ωραία αλλά τότε μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό το βέτο και η Ολλανδική κυβέρνηση ώστε να εγκρίνει ό,τι θέλει από τον προϋπολογισμό Οι Ολλανδοί και άλλοι Ευρωπαίοι λαοί όμως δεν ε, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα αυτό όπως και οι κυβερνήσεις. Περνάμε στους υπόλοιπους ομιλητές. Ο κύριος Γαρίγκα, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Λεβαντόφσκι μιλάει πάντα λογικά και γι' αυτό και η ομάδα μου τον στηρίζει. Φέτος η εντολή για τον προπολογισμό έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία από ό,τι είχε τις προηγούμενες χρονιές, δεδομένου ότι θα διαπραγματευτούμε κατά τη διάρκεια του 2012 περισσότερες δημοσιονομικές προοπτικές. Συνεπώς, η αποτυχία της εντολής στην ε, διαλογή στον τριμερή διάλογο πέρυσι που είχαμε τον Ιούνιο δημιούργησε σοβαρά προβλήματα ε, τον Νοέμβριο. Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα μπορέσουν να πετύχουν συνένεση και να τα καταφέρουν καλύτερα από ό,τι πέρυσι. Η κυρία Μπαρζάνη μίλησε για μια πολύ λογική εντολή. Περιλαμβάνονται εκεί όλες οι προϋποθέσεις οι οποίες θα μπουν σε διαπραγμάτευση για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Και επιμένει η συγγήτρια για το ότι η στρατηγική 2020 έχει πολύ μεγάλη σημασία, η ποσοτική έκφραση του προπολογισμού, για σχέδια για τα οποία δεν υπάρχουν υποχρεώσεις. Όλα αυτά θα, είναι, θα συμπεριληφθούν στον προπολογισμό 2012 και στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Η εντολή αυτή λοιπόν και ο τριμερής διάλογος θα πρέπει να προχωρήσει απρόσκοπτα. Το αποτέλεσμα τη δημοσιονομική συνδιαλλαγή του 2012 θα εξαρτηθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από τι επιτυχίε των διοργανικών διαπραγματεύσεων των επόμενων δημοσιονομικών πρακτικών. Και έπειτα έρχομαι και στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 4,9% αύξηση των πληρωμών. Ας δούμε πώς προχωράει η χρήση του προπολογισμού φέτος και τι τεράστια προβλήματα έχουμε για να γίνουν οι πληρωμές ακόμα και για το μέσο αλληλεγγύης που τόσο πολύ χρειάζεται σε πάρα πολλές περιοχές της Ευρώπης. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Καρίγα. Για 1,5 λεπτό η κυρία Γκρεγέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας και να εξάρω τη σημασία και την ποιότητα του εγγράφου αυτού για την εντολή για τον τριμερή διάλογο και που θέτει στο κέντρο των προσπαθειών μας το τη στρατηγική της Ευρώπης 2020 και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Η Κομισιόν προσπάθησε να αντιμετωπίσει την πολιτική λιτότητα των κρατών μελών αγνοώντας ουσιαστικά τη θέληση των πολιτών. Το πρόγραμμα παραγωγικά για την επιστημιστική βοήθεια για τους ε, πιο ενδεείς πολίτες είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να, <clears throat> να περικοπεί. Βλέπω από ανακοινώσεις τύπου ότι η Κομισιόν θέλει να μειώσει δραστικά το τον προϋπολογισμό που αφορά τις ε, ένα ευρώ ανακάτοικο μονάχα δίνει η Κομισιόν για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πολιτών αυτών και να υπάρξει κάποια μορφή αλληλεγγύης. Το να θυσιάζουμε λοιπόν την υποστήριξη των πολιτών αυτών στο βωμό της λιτότητας δείχνει πραγματικά ότι αστοχεί συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημασία μιας ένωσης φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους πιο φτωχούς. Δεν μπορούμε με προσχήματα τεχνικά ή νομικά να μειώνουμε την ανάγκη να υπάρξει επισητιστική βοήθεια για αυτούς οι οποίοι τη χρειάζονται. Αυτό είναι απαραίτητο για να διατηρηθεί η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραγνωρίζει τις ανάγκες των πολιτών με το να μειώνει στα τέσσερα τα ποσά τα που προέβλεπε προηγουμένως. Ελπίζω κύριε Επίτροπε ότι θα αναθεωρήσετε αυτή την απάντηση και δεν θα κοφεύσετε στους πολιτικούς στόχους και τις ανάγκες του προϋπολογισμού που εγγράφονται στο σχέδιο εντολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό. Η κυρία Γένσεν. Πούντιν. Δεν είναι παρούσα κυρία Γένσεν. Ο κύριος, ο κύριος Έλλης, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μεγάλη γυρνοδορία. Θα ήθελα να Ευχαριστώ και εγώ και να συγχαρώ την εισηγητρία. Είναι δύσκολο το έργο της υπό συνθήκες όπου προφανώς οι φιλοδοξίες της στρατηγικής του 2020 Στι οποίες συμφωνούν όλοι ότι θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν διάφορα προγράμματα και σχέδια. Ωστόσο το πρόβλημα είναι πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτές οι μεγάλες φιλοδοξίε. Υπ' αυτές τις δύσκολε συνθήκες που γνωρίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και συζητεί το Συμβούλιο. Η ομάδα μας Πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας περισσότερο στην απόδοση καλού προϊόντος από την επένδυση που κάνουμε. Όπου δεν υπάρχει καλή παραγωγικότητα θα πρέπει να περικόπτονται τα ποσά. Όπως είπε και η Επιτροπή θα είναι 0% η αύξηση των δαπανών για την διοίκηση. Ίσως θα έπρεπε να επικεντρωθούμε και σε αντίστοιχα και σε άλλους τομείς. Και έτσι να έχουμε την ευκαιρία μέχρι το φθινόπωρο να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά αυτό το ζήτημα. Έχουμε άλλωστε υποβάλει 60 ερωτήσεις σε ερωτηματολόγιο προς την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τη ζητήσουμε να εξετάσει το θέμα αυτό. Έχουμε φτάσει όμως, όπως έλεγε ένας μεγάλος κοινικός, στο να γνωρίζουμε πόσο κάνει το κάθε ένα πράγμα, χωρίς όμως να δίνουμε αξία σε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βέρτσμαν έχει το λόγο. Πρόεδρε, με το σχέδιο προπολογισμού για τον προπολογισμό 2012 πρόκειται να εξυπηρετηθούν οι στόχοι του στρατηγικής του 2020 μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Και έτσι ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια για την προσπάθειά της. Η ανάπτυξη της απασχόλησης των νέων ε, στην Ευρώπη είναι ένας μεγάλος στόχος. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά ανεργίας των νέων, μέχρι και 20% αλλά και υψηλότερα στην ε, Ισπανία. Και αυτό είναι κατανοητό γιατί στην Puerta del Sol ε, κατεβαίνουν στου δρόμου οι νέοι, όταν βλέπουμε ότι πρόκειται για μια γενιά χαμένη ουσιαστικά όπως όλοι ομολογούν. Πρέπει κάτι να γίνει για του νέου. Η στρατηγική 2020 στο σχέδιο αυτό του προπολογισμού μεταφέρει στις ε, δεσμεύσεις ε, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι στόχοι της στρατηγικής του 2020 κατά 40, περίπου 41% τα ποσά του προϋπολογισμού στις θεσμεύσει υποχρεώσεων. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Φέρμαν. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Βόν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι ότι ο υπολογισμό αφετινός και ο τριμερής διάλογος θα είναι δύσκολε υποθέσει. Ω Κοινοβούλιο λοιπόν πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για τι δικέ μα προτεραιότητες και να είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για αυτέ. Με άλλα λόγια πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κοιτάξουμε πώ θα δώσουμε πόρου για τι προτεραιότητές μα. Πρόκειται για πολιτικέ που προωθούν την απασχόληση και την ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα μάλιστα σήμερα όπου οι χώρε μέλη ε, περικόπτουν τις δικές τους τις δαπάνες. Διαφορετικά ταμεία λοιπόν για παράδειγμα, είναι πολύ βασικά για την ανάπτυξη στις περιφερειές μας. Άρα χρειάζονται την κατάλληλη χρηματοδότηση και γι' αυτό και στηρίζω την αύξηση του προπολογισμού για τα διευθυντικά ταμεία. Η έρευνα επίσης, η καινοτομία για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η έρευνα είναι πρωτής σημασίας αν θέλουμε να έχουμε απασχόληση και επιχειρήσεις. Οι επενδύσεις είναι πολύ σημαντικές επίσης στα μεταφορικά δίκτυα, στην ευρυζωνικότητα και σε περιφέρειες όπου χρειαζόμαστε περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας τώρα έχουμε νέες αρμοδιότητες και γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πρικοδοτήσουμε τις αρμοδιότητες αυτές και αυτό θέλω να ζητήσω να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Α, κύριε Επειδή φτάσατε, <clears throat> εάν θέλετε να λάβετε το λόγο, έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω να αναφερθώ στις πιστώσεις πληρωμών. Είναι πάρα πολλές χώρες οι οποίες δεν θέλουν να αυξήσουν, να δώσουν την απαραίτητη, ε, τις απαραίτητες πιστώσεις θα πρέπει να βρεθεί μια λύση και αυτή έχει να κάνει και με τις διαφορές στην ικανότητα των κρατών μελών να χρησιμοποιήσουν τα διορθωτικά ταμεία. Επιμένω ότι για τον προπολογισμό του 2012 θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια ώστε ο τομέα τη ενέργεια να αποτελέσει την προτεραιότητα. Θα πρέπει να προβλέψουμε. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα μέτρα που θα ενισχύσουν το σχέδιο για την βιώσιμη ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει επίσης το πρόβλημα του σχεδίου ΙΤΕΡ. Μας πιέζει η Κομισιόν εμάς, αλλά πρέπει να πιέσει το Συμβούλιο. Το πρόβλημα είναι στο Συμβούλιο. Εμείς υποστηρίζουμε κύριε Λεβαντόφσκι το σχέδιο ΙΤΕΡ. Ξέρετε όμως ότι δεν θέλουμε να γίνει χρηματοδότηση από άλλα ερευνητικά κονδύλια. Εκείνη το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Γένσεν. Ο κύριος Κέλλη για ένα λεπτό τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε σε γενικές γραμμές. Τα χρήματα τα οποία ε, δαπανώνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να προσθέτουν προστιθέμενη, να παρέχουν προστιθέμενη αξία και πρέπει να είναι ορατό αυτό και στους πολίτες. Αλλά η ύπαρξη προστιθέμενης αξίες και η κατάδειξη αυτή τη προσθέμενης αξία είναι κάτι το, το διαφορετικό. Πρέπει εμεί να στοιχειοθετήσουμε τέτοιο προπολογισμό που να δείχνει και στου πολίτε ότι υπάρχει προσθέμενη αξία. Επίση, η στρατηγική 2020 είναι πάρα πολύ σημαντική για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2020 θα μα κρίνουν όχι με το, με το ύψος του προπολογισμού, αλλά το αν με το αν έχουμε υλοποιήσει τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Αν υλοποιηθεί πράγματι θα έχουμε περισσότερες θέσεις ε, απασχόλησης, περισσότερη ανανεώσιμη ενέργεια, μια πιο ευφυά κοινωνία και θα είναι θετικό αυτό. Τέλο, πρέπει να τονίσω ότι χρειαζόμαστε ίδιου πόρου, Όσο νωρίτερα αποκτήσουμε αυτού του ίδιου πόρου. τόσο λιγότερο θα χρειαζόμαστε κάθε χρόνο να διαπραγματευόμαστε για τον προπολογισμό. Η κυρία Καρία άλλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα στην εισηγήτρια την κυρία Μπαρσάνη για την έκθεση που μας παρουσίασε. Πράγματι, ο προϋπολογισμός είναι το βασικό θεμέλιο που στηρίζει όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κοινή γεωργική πολιτική, την πολιτική συνοχής, έρευνας, την εξωτερική πολιτική κλπ. Δεν θα έχει κανένα νόημα Κανένα νόημα δεν θα έχουν όλε αυτέ οι πολιτικέ αν ε, δεν είχαν τη σωστή προϋποδότηση. Γι' αυτό, σε εποχή κρίση όπω είμαστε σήμερα, χρειαζόμαστε, κύριε Επίτροπε, ακόμα περισσότερο έναν δυνατό προπολογισμό ο οποίο να τα αποκρίνεται στι ανάγκε που βλέπουμε. Χρειάζονται πόροι λοιπόν για προγράμματα όπως είναι προγράμματα για την απασχόληση, την κατάρτιση των νέων ή ακόμα και για το πρόγραμμα εκείνο που έχει κόψει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις ανάγκες των πιο Επίσης λέμε στο Συμβούλιο ότι για μια φορά μη σκέφτεστε μόνο λογιστικά, για μια φορά σκεφτείτε πολιτικά και μην προσπαθείτε να βρείτε από πού θα κόψετε, γιατί θα καταλήξουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί οι πληρωμές, όπως υπενθύμησατε και εσείς κύριε Λεβαντόφσκι, είναι υποχρεώσεις νομικές που έχουμε και δεν μπορούν να περιμένουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό τώρα, ο κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Μέσα στα πάρα πολύ στενά όρια του κοινοτικού προϋπολογισμού που δεν φαίνεται ότι υπάρχει πρόθεση να, τροποποιηθεί από να τροποποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχουν δυνατότητες για ουσιαστική σύγκληση, πρέπει να κάνουμε κάποιες σημαντικές επιλογές. Και αυτό είναι απαραίτητο γιατί η μεγάλη κρίση έχει οδηγήσει σε πολύ αρνητικά αποτελέσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά συνοδεύονται με ε, απαιτήσει υπερβολικέ σε σχέση με τη συγχρηματοδότηση για τα διαρθρωτικά ταμεία. Ξέρει η Κομισιόν ποιο είναι το ποσοστό απορρόφηση των διαρθρωτικών πόρων από τι χώρε αυτέ, αλλά επιμένει να υπάρξει συγχρηματοδότηση, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα λόγω των μέτρων λιτότητο. Αυτό σημαίνει μείωση των επενδύσεων για την ερεύνα γενικά των δημοσίων επενδύσεων. Θα πρέπει λοιπόν να μειωθεί μέχρι το πολύ το 10% η εθνική συγχρηματοδότηση που απαιτείται για την ε, ε, υλοποίηση προγραμμάτων όπου υπάρχουν μεγαλύτερες δυσκολίες για να μπορέσουν τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν εκεί που είναι απαραίτητα και όχι να γυρίσουν στα ταμεία εκεί όπου δεν χρειάζεται να είναι. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αναστρέψουμε την απόκληση των οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η πολιτική του προπολογισμού έχει ένα κεφαλαιόδη ρόλο για να το πετύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μέλσεν για ένα λεπτό. Χωρίς μικρόφωνο όμως. Τώρα μ' ακούτε. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζουν όλοι ότι θα πρέπει να σφίξει το ζωνάρι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στον προπολογισμό και λόγω των εθνικών προγραμμάτων λιτότητα που θα αποτελούσε συγκρινόμενο αυτό ο προπολογισμό κόλαφο για τον πολίτη τη Ευρώπη, αλλά και γιατί είναι ανάγκη για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα προγράμματα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από του εθνικού προπολογισμού. Η μεταφορά λοιπόν κάθε χρόνο των κονδυλίων θα πρέπει των ε, πλεονασμάτων θα πρέπει να επανέρχεται στα κράτη-μέλη. Από την άλλη όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας προτείνει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση του προπολογισμού. Μπορεί οι δαπάνες για ε, διάφορα προγράμματα που ήταν πολυετή τώρα να έχουν φτάσει στην ώρα της πληρωμής. Αλλά αυτό δεν επαρκεί. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο για εξοικονόμηση πόρων και πέραν της μείωσης ε, των ποσών για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώτη ε, θέτω εγώ ως προτεραιότητα την καταπολέμηση των απατών και της διαφθοράς που θα σημαίνει πολύ σημαντική εξοικονόμηση παρόν από τον προπολογισμό. Για ένα λεπτό, κύριε Χέρτσοκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχω το χρόνο τώρα να κάνω δύο πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Η σοσιαλιστική ομάδα <clears throat> υποστηρίζει τη δημιουργία του του ΙΤΕΡ <clears throat> δεν συμφωνεί όμως με την μεταφορά 100 εκατομμυρίων ευρώ από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Θα θέλαμε επίσης τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και τα προγράμματα για την διαδικτύωση της ενέργειας να έχουν και μια ευελιξία κατά 5%. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευελιξία γιατί είναι μια προϋπόθεση για το να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει προς τον τομέα της ανάπτυξης. Ευχαριστώ την κυρία Έρτσοκ. Δίνω το λόγο τώρα στον Επίτροπο Λεβαντόφσκι. Yes. remark, anticipating. Σύντομα και πριν από τον τριμερή διάλογο. Θέλω να απαντήσω σε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ο κύριος Καπούλας Σάντος αλλά και η κυρία Γκρελιέ υποστηρίζουν το πρόγραμμα για τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πώς αντέδρασε όσον αφορά τα πλεονάσματα που θέλουμε να πάνε στους πιο ευάλωτους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βρούμε μία λύση και να βρούμε κατά πάσα πιθανότητα μια νέα νομική βάση. Η δεύτερη σύντομη παρατήρησή μου προς τον κύριο Πατικόφερ. Είπατε ότι δεν φαίνονται καθαρά προτεραιότητά μας για την ενεργειακή πολιτική εξαιτία της υποχρηματοδότησης. Φέτος όμως, εξαιτία της καθυστέρησης προγραμμάτων επενδυτικών του Ναμπούκο, για παράδειγμα, και άλλων, για το Αζερβαϊτζάν, κέρδισε τη Eurovision το Αζερβαϊτζάν. Και έτσι Καθυστερήσαμε πολύ. Και όσον αφορά τις ενεργειακές διασυνδέσεις. Όσοι λοιπόν θέλουν περικοπές στον προπολογισμό, πρέπει να τους πω ότι βάσει των νομικών υποχρεώσεων που έχουμε το 2012 πρέπει να πληρώσουμε και την Ελλάδα και άλλες χώρες που έχουν δυσκολίες. Χρειάζεται λιτότητα, αλλά χρειάζονται και επενδύσεις. Οι νομικές μας υποχρεώσεις είναι ε, πάνω από τις επενδύσεις για τις χώρες αυτές για τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε η κυρία Μπαλτζάνη τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από αυτή την τόσο σημαντική και ενδιαφέρουσα συζήτηση και από αυτές που κάναμε στις ε, επιμέρους Αρμόδιε επιτροπές φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη σύμπνοια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε. Μεταξύ των πιο σημαντικών στοιχείων. Ο προϋπολογισμός είναι προφανώς το μοναδικό ή και το πιο σημαντικό στοιχείο για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τις ισορροπίες μεταξύ της λιτότητας των δημοσίων λογαριασμών και της ανάγκης να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη. Είναι το μόνο, ο μόνος προμαχώνας που έχουμε εναντίον της ύφεση η οποία μπορεί να προκύψει από την ε, παγιοποίηση των εθνικών προϋπολογισμών. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ζητάει ένα φιλόδοξο προϋπολογισμό. Ζητάει όμως να υπάρξει ένα εργαλείο ισχυρό το οποίο θα ενισχύσει τις προτεραιότητες οι οποίες είναι ορατές και αναγνώσιμες. Η στρατηγική του 2020 απαιτεί επενδύσεις για την δημιουργία θέσεων εργασίας. Έχουμε τονίσει τη σημασία της έρευνας, της ενέργειας, της κοινωνικής συνοχής. Όλες αυτές είναι προτεραιότητες για τις οποίες σήμερα η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό θα είναι και η λιδία λίθος της ε, αξιοπιστίας και της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, σήμερα παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο προϋπολογισμός γιατί πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι αυτό θα είναι και ο μοχλό, θα είναι η κινητήρια δύναμη η οποία θα μπορέσει να βοηθήσει οι οικονομίε μας να ξεκινήσουμε. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν μπορούμε να εξασφαλίσουμε να επαναφέρουμε την σταθερότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και του ενιαίου νομίσματός μας. Νομίζω ότι ήδη μέσα σε αυτό το τριγωνικό διάλογο, μέσα σε ένα πνεύμα υψηλής ευθύνης γιατί δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, θα πρέπει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις γαλήνιες, υπεύθυνε και επικοδομητικές για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπαλτσάνη. Έχει κλείσει λοιπόν αυτή η συζήτηση. Στις 12 σήμερα θα ψηφίσουμε και περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι η κοινή συζήτηση για την πολιτική συνοχή. Και έχει καταρχήν το λόγο για 4 λεπτά κύριος Πίπα.